Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ξεκινούμε με το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, απαλλαγή του προϋπολογισμού. Ανδρέα Τσέσκοβα, η συγγήτρια. Και να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στην κυρία Τσέσκοβα. Vážený pane není to co se tady Συνάδελφοι, δεν είναι πρώτη φορά που συναντιόμαστε για να συζητήσουμε σχετικά με το ίδιο σέμα. Με ακούτε, μεταφράζομαι. Děkuji. Ε, setkáváme Όχι, δεν είναι πρώτη φορά. o udělení. Που συζητάμε αυτά τα σχετικά με το δεύτερο σχέδιο κειμένου της ε, έκθεσης που αφορά την απαλλαγή ε, για το Συμβούλιο για τη χρήση του 2011. Όπως τα ξέρουν όλοι οι συναδέλφοι, κατά τις χρήσεις του 9 αλλά και του 10 είχαμε μια κατάσταση ταυτόσιμη. Οπότε και σύμφωνα με την, ε, είχαμε την έκθεση που κατέληξε σε απέρριψη, σε απόρριψη. Οπότε να μην σας πω όλες τις ε, λεπτομέρειες, αλλά πάντως όπως και για τις προηγούμενες χρήσεις το Συμβούλιο απεφάσισε να μην υποβάλει τις παρατηρήσεις που ζητήσαμε. Ίσως τα θυμάστε. Η Επιτροπή μας είχε υποβάλει 52 ερωτήσεις στο Συμβούλιο σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά το Συμβούλιο. Αυτά για τη χρήση 2011 δεν απήντησαν. Δεν άλλαξε τίποτα από τότε σε σχέση με τα δύο προηγούμενα οικονομικά αιτία. Συνήθισα προσωπικά εκπροσώπους της Βελγικής Προεδρίας. σε ενημέρωση, είπαμε ότι έχουμε δύο ερμηνείς που επιδέχεται το σχετικό άρθρο της ε, συνθήκης όσον αφορά την ενημέρωση του Συμβουλίου προς το Κοινοβούλιο. Ε, υποστηρίζεται κατά τη μία ερμηνεία ότι το Συμβούλιο δεν υποχρεούται να υπόκειται σε έλεγχο των χρηματοοικονομικών του από το Κοινοβούλιο, όπως υποχρεούνται τα άλλα θεσμικά όργανα. Άρα ε, αυτό έχει συνέπειες και όσον αφορά την απαλλαγή. Αυτή την ερμηνεία του το Συμβούλιο, σε αυτήν εμένη, όπως και στο προηγούμενο δεν άλλαξε τίποτα και, εν πάση δεν έχω κάποια πάλι πληροφορία, κάποια άλλη ενημέρωση ότι μετέβαλε την τοποθετησή του το Συμβούλιο. Παρά την αλλαγή της Προεδρίας. Δεν ξέρω τώρα μήπως και η Λιθουανική Προεδρία προσεγγίσει διαφορετικά το ζήτημα αλλά πάντως προς το παρόν δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Τα ίδια όπως πέρυσι και πρόπερσι. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, σε αυτό το κλίμα, σύνταξα το κείμενό μου, οπότε για άλλη μια φορά θα αρνηθούμε την απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Βέβαια, η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου αλλά και το εργαστήριο το εργαστήριο το οποίο συγκροτήσαμε πέρσι για το θέμα αυτό έχουν τοποθετηθεί. Λένε ότι το δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο που είναι το Κοινοβούλιο είναι υπόλογο προς τους Ευρωπαίους. Άρα και γι' αυτό έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα επί του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών. Έχουμε επομένω εδώ πέρα δύο αντικρώμενε ερμηνείε του νόμου. Πώς θα έρθει τώρα αυτή η αντίφαση. Ο μόνος τρόπος είναι να γίνει διάλογος με την Προεδρία. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε εξελίξεις προς το καλύτερο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ό,τι παρατηρήσεις, σχόλια έχετε, ευπρόσδεκτο. Περιμένω τις τροπολογίες σας επίσης. Ευχαριστώ, κυρία Τσέσκοβα. Λοιπόν, Υπάρχουν σχόλια. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο για τα όσα είπε η κυρία Τσέσκοβα. Ο κύριος Βαλτσίτης και μετά ο Γιάννη Μούλτερ. Πρώτα ο Σιγμάντας. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Για τρία χρόνια, τρία χρόνια το ακούμε αυτό το πράγμα και είναι λογικό και για όλους μας είναι σαφές ότι ότι ανεξάρτητα όταν έχουμε δημοσιονομική αρχή, η αρχή πρέπει να ακούει τη λογοδοσία του Κοινοβούλιο. Αυτό ωστόσο γίνεται πια πολιτικό θέμα, δεν είναι μόνο οικονομικό ή πολιτικό η Προεδρία της Λιθουανίας ή οποιοδήποτε άλλο κράτος δεν μπορεί να το λύσει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των οργάνων της Ένωσης. Τι αν δεν δώσουμε απαλλαγή για τρίτη συνεχή φορά θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια μέτρα. Άλλο δρόμο δεν βλέπω. Αλλιώς δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν αν τα χρήματα ξοδεύονται σωστά. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Γιάν ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ε, πάντα το ίδιο κάνουμε κάθε χρόνο και μπορούμε να το κάνουμε και φέτος και μπορούμε να το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ίσως καλό να είναι και αυτό που λέει η συγκήτρια, να προσπαθήσουμε και πάλι να έρθουμε σε επαφή με τη Λιθουανική Προεδρία. Να τους καλέσουμε εδώ, για να μας πούνε την άποψή τους. Και το θέμα είναι, θέλουμε να κάνουμε ό,τι κάνουν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα ή είναι τόσο πια ιδιαίτερη περίπτωση στο Συμβούλιο που δεν θέλουμε. Αυτά. Ε, άλλοι δύο συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Ο Σόρεν πρώτα και μετά ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για το σχέδιο. Συμφωνώ. Πρόκειται για καλή, για καλό σχέδιο. Επίσης, συμφωνώ με όσους λένε ότι δεν μπορούμε να αναβάλουμε μάλλον δεν μπορούμε να μεμφθούμε την Λιθουανική Προεδρία. Το Συμβούλιο είναι αυτό που φταίει. Η Λιθουανία είναι μια μικρή χώρα, νέα χώρα, σχετικά νέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ δύσκολα νομίζω θα μπορέσει να κινήσει τα πράγματα στο Συμβούλιο. Η συγκατάσταση στο Συμβούλιο είναι αυτή που είναι εδώ και χρόνια. Τι να κάνει και μια έρμη λιθωνική προεδρία. Θα ήταν σκόσπιμο τόσο παρά τα αυτά να μιλήσουμε με τους εκπροσώπους της Προεδρίας και θα πρέπει να τους εκλυπαρίσουμε να ακολουθήσουν αυτά που είχε κάνει η Σουηδική Προεδρία. Δεν είναι όλες οι προεδρίες οι ίδιες. Θυμάμαι ότι υπήρχε μία προεδρία, η Δανέζη για παράδειγμα, που ε, δεν μας έδωσε τίποτα. Αλλά υπάρχουν και διαφορετικές. Σουηδία, γειτονική χώρα σε μένα, που έδωσε έμεσα μεν απαντήσεις δε σε ορισμένα ερωτήματά μας. γραπτές απαντήσεις μερικές φορές στη, ε, στο site της Προεδρίας όπου έλεγε το κοινοβούλιο μας ρώτησε αυτό και εμείς θα απαντήσουμε αυτό κάτι έμεσο τέλος πάντων να θα μπορούσαμε να πούμε στους Λιθουανούς μιμηθείτε τους ε, Σουηδούς μη μιμηθείτε τους Δανούς δεν είναι οριστική λύση αλλά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση Ευχαριστώ πολύ, Σόρεν. Ο κύριος Αντί. Merci, Monsieur le Président. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Και ευχαριστώ την συντονίστρια. Ποτέ δεν συμφώνησα με την τεχνική επιλογή της Επιτροπής, γιατί το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι το Συμβούλιο δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση που έχει την πολιτική και δημοκρατική, ούτω ώστε να παράσχει ό,τι στοιχεί στη διάθεσή του στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να ασχίσουμε την ελεκτική μα αρμοδιότητα, την δημιουργική αλλά και πολιτική επί τη εκτελεστική εξουσία. Άκουσα προσεκτικά πάντως το θέμα, άκουσα για τις δύο διαφορετικές ερμηνείες. Ε, νομίζω τα πράγματα έφτασαν στα άκρα. Αδιέξοδο. Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση για την απαλλαγή. Αλλά η ανάλυση αυτή είναι λανθασμένη γιατί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η της Λισαγόνας υπάρχει ενιαία νομική προσωπικότητα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελεστική εξουσία είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη μεριά έχουμε ε, τα υπόλοιπα όργανα, το Συμβούλιο, Ελληνικό Συνέδριο κλπ. Και η παράδοση είναι παλαιότερη όσον αφορά την απαλλαγή και λαμβάνει υπόψη ε, αυτή η παράδοση τα καινούργια στοιχεία, δηλαδή αυτήν την ενιαία νομική προσωπικότητα της Ένωσης. Δεν έχουμε αρμοδιότητα, ε, λένε. Ε, όχι, έχουμε. Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τους λογαριασμούς, τα χρηματοοικονομικά όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το λίγο συνέδριο που έχει την ελληνική αρμοδιότητα, ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ λίγε ε, παρατηρήσει προ το Συμβούλιο. Αυτό είναι λίγο παράδοξο. Γιατί έχουμε αυτέ τι 200 σελίδε. Ε, αλλού και δίνουμε την απαλλαγή. Ενώ εδώ πέρα έχουμε ελληνικού συνεδρίου πέντε παρατηρήσεις και την αρνούμεθα. Επομένω είναι απαράδεκτο το να μην παρέχει την ενημέρωση που πρέπει το Συμβούλιο. Απαράδεκτο. Και απαράδεκτο δεν πάει να πει ότι ε, φταίει ο πρόεδρος της Λιθουανίας της Ιρλανδίας. Φταίνε οι υπάλληλοι του Συμβουλίου. Αυτοί έχουν αυτή την πολιτική. Αυτοί βρίσκονται ένα δίκο και δεν δίνουν στους εισηγητές μας τις πληροφορίες που χρειάζονται. Τα πράγματα όμως έχουν περιπλάκει τώρα και υπηρεσία. Εξωτερικές δράσεις παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί να μην δώσουμε την απαλλαγή. Είναι μια αντότητα. Και λέμε Έχουμε συμβούλιο, από έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι μια οντότητα ταυτόσιμη, ολόιδια, ίσως όσον αφορά τη διοικητική λειτουργία. Τέλο εγώ δεν έχω τη λύση, αλλά θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και αναρωτιέμαι, μήπως η λύση θα ήταν να εμπλέξουμε εδώ τους ε, φίλους εθνικούς βουλευτές να γίνει κάποια κινητοποίηση προς τα εκεί, μέσω του Πρόεδρου του Κοινοβούλου και ίσως όλοι οι πρόεδροι των Επιτροπών Δημοσιονομικού Ελέγχου των Εθνικών Κοινοβουλίων που ελέγχουν ε, τα κράτη τα οποία συμμετέχουν στο Συμβούλιο να πούνε κοιτάξτε ε, οι υπάλληλοι του Συμβουλίου δεν παρέχουν τα σχετικά έγγραφα εάν τελικά προκύψει ότι υπάρχουν κάποιες ιεραρχικές εντολές από πλευράς Προεδρείου ή Υπουργών Προεδρίας, τότε το πρόβλημα είναι πραγματικά πολιτικό. Οπότε, Πρόεδρε, θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε κάτι σαν ατομική βόμβα. Γιατί όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει την εκτελεστική εξουσία που είναι υπεύθυνη ενώπιόν μας και από πλευράς δίνησης του ελέγχου και από πλευράς πολιτικής είναι υπεύθυνη. Οπότε θα ρίξουμε την ατομική βόμβα, αυτή την απειλή της βόμβας που θα είναι απειλή ε, μεγάλης εμβέλειας. Αλλά προσοχή να μην κάνουμε κάτι που να είναι δυσανάλογο, πολύ δυσανάλογο. συνομιλημένος από την Ιστονίστρια και από τους συναδέλφους ακριβώς γιατί διαχωρίζω τη θέση μου, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί το Συμβούλιο στην Ολομέλεια, γιατί παίζει αυτό το ηλίθιο παιχνιδάκι. Και τελικά οι ευρωσκεπτικιστές πρόκειται να ωφεληθούν. Θα πει να δώστε τα οδηπορικά, ε, αποκαλύψτε τα, τις δαπάνες σας, ε, δώστε την απαλλαγή, αλλά μιλήστε με τον μα. Δεν είναι αυτό συμπεριφορά εντάξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν από νομικέ πλευρά δεν μπορέσουμε να επισημάνουμε ποιε είναι οι σωστέ αρμοδιότητε, ε, τότε ας καταφέρουμε με τη σωστή συμπεριφορά να δώσουμε την απαλλαγή. Αλλιώ ε, γελιοποιούμε εμεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Οντή για την ε, λαμπρή αναφορά σα. Κυρία Γκρέσλε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να θυμίσω ότι πολλές φορές έχουμε κάνει συζητήσεις για το κατά πόσο η Γαλλία είναι δημοκρατία. Να θυμίσω στον κύριο Ντί. Πάντα εγώ τη θέτω αυτή την ερώτηση, το παραδέχομαι. Γιατί αν κοίταξει κανείς το Σύνταγμα, ε, κάποια πράγματα μπορεί να το αφισβητήσει. Εν πάση περιπτώσει. Ε, πρέπει να πω ότι Έχουμε κάθε λόγο να μην δώσουμε την απαλλαγή στο ε, Συμβούλιο και δεν ε, είναι σωστά αυτά που λέγονται υπέρ της απαλλαγής. Καταρχάς, το ελεκτικό συνέδριο. Αν δούμε τι έχει κάνει, το, έχει εξετάσει το ελεκτικό συνέδριο τον τίτλο 5, θα πρέπει να παρακαλέσουμε τους εκπροσώπους να μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες που έχουν για το πόσες πληρωμές έχει εξετάσει το ελεκτικό συνέδριο από τον προπολογισμό του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει καμία παρατήρηση στον, ε, στον προπολογισμό του Συμβουλίου. Όχι γιατί δεν έχουν γίνει, ε, όχι γιατί είναι όλα σωστά τα στοιχεία, αλλά γιατί δεν έχουν γίνει ε, οι έλεγχοι. Πρέπει να, να εξεταστούν οι πληρωμέ σε όλα τα, σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, σε όλες τις υπηρεσίες. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Ε, θα μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος δεν άλλαξε. Το Συμβούλιο μας ε, ε, δίνει, μας κουνάει ένα χαρτί μπροστά μας όπου είναι 20 χρονών χαρτί. το κάθε θεσμικό όργανο έχει τη δική του ευθύνη για το δικό του προπολογισμό. Ή το 235 είναι ή το 335 άρθρο αυτό. Οπότε Μπορούμε να κάνουμε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε πουθενά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και νομίζω ότι θα είναι σωστό, είναι να, να τηρήσουμε την στάση που έχουμε τηρήσει. Ε, εντάξει, θα, ε, δεν θα δώσουμε την ε, δεν θα δώσουμε την ε, απαλλαγή στο, κοινοβούλιο, στον ε, Συμβούλιο συγγνώμη, για τέταρτη χρονιά και τι έγινε. Στην Κομισιόν πόσες φορές έχουμε ζητήσει να μας δείξει την ε, σχετική δήλωση. 20 φορές την έχουμε ζητήσει και δεν έχουμε λάβει ποτέ. Λοιπόν, στα διάφορα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκαν τώρα, πρόσφατα με πάση περιπτώσει, έχουμε, κάνει διαφορετική, έχουμε ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία. Δεν, τι, δεν κάναμε την ίδια, δεν είχαμε την ίδια μεταχείριση. Γι' αυτό, Ζαμπιέρ, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Το Συμβούλιο, εντάξει, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι άλλο. Είναι, ο προπολογισμό του είναι δικό του. Αλλά θα πρέπει στο τέλο να σκεφτούμε αν όντως όλα αυτά θεωρούνται κομμάτια της Κομισιόν με 10 διαφορετικούς επιμέρους προπολογισμού, ε, τους οποίους κάθε φορά πρέπει να εγκρίνει η Κομισιόν. Α λάβουμε ίσω ε, τι πληροφορίε από την Κομισιόν για το Συμβούλιο. Αλλά τέλο πάντων αυτό είναι γραφειοκρατία. Εμεί ρωτάμε την Κομισιόν, η Κομισιόν ρωτάει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο βεβαίω ε, θα προσπαθήσει εμέσω να απαντήσει την Κομισιόν και μετά μέσω των τριών αυτών ε, θεσμικών οργάνων να καταλήξουμε εμεί να πάρουμε τι πληροφορίε μα. Ε, δεν μπορούμε τώρα να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε και το μέσο που έχουμε είναι ο προπολογισμό. Ερώτημα λοιπόν, αυτή η συμφωνία κυρίων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την απαλλαγή δεν θα πρέπει να την τηρήσουμε, να την τιμήσουμε. Αλλιώς να τη διαγράψουμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας. Νομίζω ότι όλοι τώρα ε, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τον πιο εύκολο δρόμο. Νομίζω ότι θα κάνουμε λάθος να φύγουμε από την θέση μας, να παρεκκλίνουμε από τη θέση μας. Ε, θα μπορούσαμε και τα επόμενα χρόνια να μην δώσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Πολύ, ε, εγώ ευχαριστώ. Όντως πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση για την άρνηση της απαλλαγής στο Συμβούλιο. Εντάξει, περάσαμε και σε πιο φιλοσοφικά θέματα όπω το αν η Γαλλία είναι δημοκρατία, αλλά ε, είναι κάνει και ζέστη. Είναι και Ιούλιος. Όχι, όχι, Ίγκε. Ε, πρόεδρε. Ε, ναι, αλλά τώρα αν γελιοποιείς αυτά που λέω... Ε, εντάξει, ίσως είναι λίγο προσωπική η κόντρα ε, για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Τώρα εντάξει, για να συζητήσουμε για το αν η Γαλλία είναι δημοκρατία ή όχι είναι άλλο θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατική παράδοση στην κάθε χώρα είναι διαφορετική. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Κοινοβούλιο δεν αποφασίζει για, μια, για τις δαπάνες της κυβέρνησης. Δεν μπορώ καν να το φανταστώ. Εντάξει, πριν πάρει ο Ζαν Πιεροντή λοιπόν το λόγο, να πω ότι για τις διάφορες παρα... δημοκρατικές παραδόσεις ε, των διαφόρων χωρών, εγώ σκέφτηκα κατευθείαν την Ουγγαρία για κάποιο λόγο. Λοιπόν, Ζαν Πιέρ, εντάξει, αν ξεκινήσουμε τώρα τούτη τη συζήτηση, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Λοιπόν, Ζαν Πιέρ. Να σας επιβεβαιώσω ότι η Ουγγαρία είναι δημοκρατική χώρα, αλλιώς δεν θα ήταν μέλος της Ένωσης. Μη φοβάστε λοιπόν, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι έχουμε θετικές ανταλλαγές για τους μεν και για τους δε. Also, das Ωραία. Θα το γράψουμε στα πρακτικά. Εντάξει. Μας καθησυχάσατε. Άλλος κανείς. Όχι. Ωραία. Η συγγήτρια, αν θέλει, και πάλι να πάρει το λόγο. Κυρία Τσέσκοβα, θέλετε να μιλήσετε και πάλι για να κλείσουμε, αν θέλετε. Ναι. Να πω δύο λόγια κι εγώ. Διασκεδαστική ήταν η συζήτηση νομίζω. Τέλος πάντων, θέλω να σας ευχαριστήσω πιο σοβαρά τώρα για τα πολλά σχόλια που κάνατε. Βλέπω ότι μπορούμε να δουλέψουμε με νέο τρόπο. Δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ μας και να απαντήσω σε κάποια σχόλια. Ναι, το θέμα έγινε πολιτικό. Καλό είναι αυτό. Γιατί αν το δούμε από την νομική άποψη, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες της συνθήκης. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πολιτική άποψη που σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε έναν διάλογο. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν δύο πλευρές που θα μετέχουν στο διάλογο και που θα θέλουν να συνεργαστούν. Και αυτό ζήτησαν οι περισσότεροι συνάδελφοι, ζητώντα από το Συμβούλιο να δείξει βούληση συνεργασίας. Αναφέρθηκε ήδη ότι πρέπει να καλέσουμε έναν εκπρόσωπο τη προεδρία. Δεν μας εμποδίζει κανεί να το κάνουμε αυτό. Βεβαίω εξαρτάται από την, την ηγεσία τη επιτροπή μα. Εγώ θα ήμουν υπέρ τη πρόταση. Κάτι άλλο που τέθηκε στη συζήτηση. Η Προεδρία δεν θα μπορέσει μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει την πορεία που έθεσαν οι προηγούμενες Προεδρίες. Συμφωνώ ωστόσο ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και το Κοινοβούλιο όντως είναι δημοκρατικό όργανο. Και να εξηγήσουμε γιατί μιλάμε για δεύτερη έκθεση, αλλά μιλάμε για την απαλλαγή του οικονομικού έτους 2011. Υποθέτω ότι τα επόμενα έτη θα υπάρχουν δύο εκθέσεις για τα δύο θεσμικά όργανα σε σχέση με τη νέα κατανομή. Μία για το Συμβούλιο, μία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό προς το παρόν, παρότι μου ζητήθηκε στην αρχή να ετοιμάσω δύο εκθέσεις. Μία τελευταία παρατήρηση. Βάσει της συνθήκης, όντως, θα έπρεπε να δώσουμε την απαλλαγή στην Επιτροπή, που είναι υπεύθυνη και λογοδοτή για την εφαρμογή των ετησίων λογαριασμών. Αλλά αυτό στηρίζεται στην έρχεται σε αντίθεση με την ε, άρνησή τους να μας επιτρέψουν να ελέγξουμε τους λογαριασμούς του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι είναι σαφές από την έκθεση ότι το Κοινοβούλιο ως δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο έχει αυτό το δικαίωμα ότι πρέπει να μπορεί να δεχθεί το γεγονός αυτό και να ξεκινήσει ένα διάλογο. Βέβαια, αν δεν υπάρχει σαφής ερμηνεία της συνθήκης, συνεχίζουμε τις συζητήσεις. Διότι αυτό, πάνω σε αυτό, έχει στηριχθεί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το διάλογο και τη συζήτηση. Πάντως δεν είναι λάθος της Επιτροπής μας ή του Κοινοβουλίου. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με την άλλη πλευρά. Θέλω να ευχαριστήσω και τη, γραμμα... και τη Γραμματεία για τη συνεργασία. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Πιστεύω ότι η συζήτηση έδειξε πως θα έπρεπε να αρνηθούμε την απαραγή. Δεν βλέπω άλλη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Τσέσκοβα. Να πω ότι οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2013 στις 12. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό. Το σημείο 8. Πάμε στο σημείο 10. Το 9 είπαμε ότι ακυρώθηκε. Πάμε στην ειδική, επιτροπή, στην ειδική έκθεση 21-2012 το αποτελεσματικότητα προς το κόστος της πολιτικής συνοχής και των σχετικών επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. Ο κύριος Μπαλτσίτης είναι ο εισηγητής. Να του δώσουμε λοιπόν το λόγο για κάποια εισαγωγικά σχόλια. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βίγκα Μπάουερ για από το ε, ελεγκτικό συνέδριο. Ο Ζιγμάντας έχει το λόγο. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami kolegos. Jau mes aptarėme pačio dokumento esmę šiek tiek anksčiau. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήδη συζητήσαμε το κείμενο. Οπότε με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το ελληνικό συνέδριο. Μα επικρίνουν, αλλά το έγγραφο είναι πολύ αξιόλογο. Επίση, να ευχαριστήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και επίσης έγινε αντιληπτό το πρόβλημα. Δεν υπήρξε καμία απόπειρα συγκάλυψη Οπότε, και έχουμε κάποια συγκεκριμένα ε, βήματα που πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε και τη γραμματεία να ευχαριστήσουμε γιατί βοήθησαν για την έκθεση. Όπως είπαμε, αυτή η έκθεση καλύπτει την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση. Τσεχία, Λιθουανία, οι προγράμματα που τρέχουν από το 2000 μέχρι το 2013, οπότε έχουμε τρία προγράμματα τα οποία καλύπτουν την περίοδο αυτή, 2007-2013 ε, και έχουμε και ένα 2000 με 2006. Στην έκθεσή μου Συνεφώνησα καταρχήν με τα συμπεράσματα του Ελληνικού Συνεδρίου. Η αποδοτικότητα δεν ήταν εξαιρετική. Αλλά δεν είχαν ταχθεί και κάποιοι κανόνες, κάποια πρότυπα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάπως περίπλοκο σήμερα, αναδρομικά δηλαδή, να ε, ε, εγκρίνουμε, να, αποτιμήσουμε σε τα προγράμματα. Η νέα οδηγία για την ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2014. και πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσει γιατί δεν έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Να υπόψη όλα όσα είπε η Επιτροπή αλλά και το Ελληνικό Συνέδριο. Ιδίω εκεί που λέει για συγκεκριμένου δείκτε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 14 με 20 ανάλυση των επιπτώσεων, η υποχρεωτική έλεγχη για την ενέργεια, ό,τι δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Και τώρα η αξιολόγηση της ε, αποκτικότητας των μέτρων για την ε, πολιτική ενεργής απόδοσης θα γίνει μέσα σε λίγα χρόνια. Ε, επίσης είπαμε ότι τονίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν κριτήρια επιλογή Αυτό αφορά και του διαγωνισμού τις προμήθειες και όσου διαγωνισμού γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτά πιστεύω θα βοηθήσουν. Ό,τι παρατηρήσει έχετε, πρόσδεκτε. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπαλτσίτης, να δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ευτυχώς ε, έχουμε κάνει την ενδιαφέρουσα συζήτηση ήδη μια φορά, την οποία κλείσατε με πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρατηρήσεις για τις οποίες θέλω να σας ευχαριστήσω. Ε, ε, σύντομα λοιπόν, μια σύνοψη θα κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτή η έκθεση έχει συζητηθεί πάρα πολύ εντατικά, όχι μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει, είχαμε κάνει και μια συζήτηση περίπου μια μισή ώρα και στο Συμβούλιο. Ε, δεν είναι συχνό το φαινόμενο να συζητούνται τα, οι ειδικέ αυτέ εκθέσει στο Συμβούλιο. Και μετά από αυτή τη συζήτηση λοιπόν στο Συμβούλιο έγιναν κάποιες, λήφθησαν κάποιε αποφάσει για την σύναψη συμπερασμάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ πολύ λοιπόν για την έκθεση αυτή. Τώρα, ε, σε σχέση με, το, με τα όσα περιλαμβάνει η έκθεση, ε, περιλαμβάνει απολύτω τις προθέσεις μας και θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν γιατί η Κομισιόν δραστηριοποιήθηκε ήδη τον Απρίλη είχε δραστηριοποιηθεί, είχε υποβάλει νέες προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Και ο τομέας αυτός, όπως είπε και ο κύριος εισηγητής, είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για το, για το στόχο 2020. Αν λοιπόν συνεχίσουμε έτσι όπως είχαμε κάνει μέχρι τώρα, να έχουμε δηλαδή ένα περίπου 10 έως 20% των μέσων για την, ε, να πηγαίνουν στην ενεργειακή απόδοση, ε, θα, έχουν, θα έχουμε ε, δυσκολίες στο να πετύχουμε τον στόχο για τον άνθρακα στο πλαίσιο του 2020 Χαίρομαι λοιπόν που η Κομισιόν το υποστηρίζει και ξέρει ότι αυτό πια είναι στόχος της πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και το Κοινοβούλιο βεβαίως, αλλά και την Κομισιόν. Και όπως είπε και ο εισηγητής, το πιο σημαντικό είναι ότι θα δούμε στο μέλλον εάν αυτές οι καλές ε, αποφάσεις που πήραμε ε, δουλεύουν. Εμείς ευχαρίστως να βοηθήσουμε και στο follow-up και επίσης μπορώ να σας ανακοινώσω ότι προς το παρόν τρέχει μία έκθεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτή η έκθεση θα ολοκληρωθεί σε λίγο καιρό. Βλέπετε ότι ε, ακριβώς ε, πάνω σε αυτό το ζήτημα, πάνω σε αυτό το τομέα, ε, ε, δραστηριοποιούμεθα και εμείς περαιτέρω. Επίσης για την, κλιματική, για την προστασία του κλίματος θα υποβάλουμε μια νέα έκθεση. Μπορείτε λοιπόν να βασιστείτε πάνω μας για τον τομέα αυτό. Ξέρουμε ότι είναι πολιτικά πολύ σημαντικός τομέας. Δεν είμαστε μόνο ελεγκτικό συνέδριο, αλλά και εμείς σκεφτόμαστε πολιτικά και γι' αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και εσά και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, έτσι ώστε να επιτύχει του στόχου της. Αλλά ε, όπως είπαμε, όταν δοκιμάζει κανείς ε, το γλυκό βλέπει αν το έκανε καλά. Γι' αυτό ε, πρέπει να περιμένουμε δύο-τρία χρόνια για να δούμε αν όντω τα μέτρα που παίρνουμε τώρα έχουν τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρατηρήσεις υπάρχουνε. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ναι. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου γιατί η ενεργειακή απόδοση είναι πραγματικά προτεραιότητα ευρωπαϊκή και έχουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες ό,τι αφορά και την πολιτική απασχόληση για τα μέτρα της, μέσω των μέτρων των, της ενεργειακής απόδοσης, για τα για τα έξυπνα κτίρια και αυτό βεβαίω θα καταστήσει και την ενέργεια πιο φτηνή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων για του πολίτε μα. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξή. Το ελεκτικό συνέδριο βλέπει αν υπάρχουν κάποιε συνέπειε και σε ό,τι αφορά την απασχόληση μέσω του προγράμματο. Και επίση, ποιε προοπτικέ υπάρχουν στην Ευρώπη, 1,2 εκατομμύρια σπίτια πρέπει να βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση. Οπότε υπάρχει ε, ένας τεράστιος όγκος εργασίας εδώ και σε διαφορά τα παράθυρα, τι ε, τις μονώσεις, ε, τις στέγες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία θέσεων εργασίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η έκθεση αυτή να τύχει της δέουσης προσοχής και από εμάς. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι μάλλον. Οπότε ε, ο εκπρόσωπο του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου. Ναι, να απαντήσω. Βεβαίω είναι εντατικό ο τομέα αυτό ω προ την απασχόληση και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δομηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι όπως το κάνουν διάφορες χώρες. Δηλαδή, να έχουμε μία ε, απόδοση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις μας. Έχουμε για περίπου 150 χρόνια, ένα όριο 150 χρόνων για απόσβεση των των επενδύσεων, αλλά αυτό δεν φέρνει θέσει εργασία. Θέσει εργασία φέρνουν αυτά που είπε ο ε, κύριο Ευρωβουλευτή. Ε, Επενδύσει ε, στου σωστού τομεί και όπω αναφέρθηκε και στην έκθεση του δική μα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Πρέπει να καθοριστούν, ε, πρέπει να καθοριστεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απόσβεση, ε, ένα κέρδο από τούτη την επένδυση. Ακόμα και από τι μικρέ επενδύσει για τα νοικοκυριά, ας πούμε, είναι διαφορετικές οι επενδύσεις και διαφορετικό το, το κέρδος που έχουμε από αυτές και είναι διαφορετικές οι επενδύσεις και το κέρδος στον δημόσιο τομέα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας, έτσι με, δύο, ε, με ένα σβάρο δύο τριγώνια μπορούμε να έχουμε και ε, δημιουργία θέσεων και ενεργειακή απόδοση. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε εκεί που μπορούμε να εξοικονομήσουμε και ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα. Είναι λοιπόν αρκετά θετικό γιατί όντως μπορούμε και να, μειώσουμε, και να ε, μειώσουμε την ενέργεια και να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Ωραία. Να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν λοιπόν. Θέλετε να απαντήσετε, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Κόπενς έχει το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλτσίτης που ανέλαβε, που έλαβε υπόψη της απόψης Επιτροπής ε, στην τελική του σύσταση και να τον ευχαριστήσουμε και για την έκθεση. Πολύ σημαντική έκθεση για μας, μας διαβεβαιώσω ότι αν δείτε την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, οι επενδύσει στα μέτρα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα τη ενέργεια θα αποτελέσουν προτεραιότητα στα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα των Και όπω γνωρίζετε καλά, τούτο αντικατοπτρίζεται και στη θέση της Επιτροπής για τα προγράμματα αυτά μέσω των ε, position paper που έχουμε και θα προσπαθήσουμε τα ευρήματα της έκθεσης να δώσουν αποτελέσματα. Κάποια σχόλια που θέλω να επαναλάβω. Πρώτον, το κόστος επένδυσης ανά την Ένωση είναι δύσκολο να εντοπιστεί λόγω του ότι υπάρχουν διαφορετική τιμολόγηση υλικών, ε, ε, εξοπλισμού και προφανώς υπάρχουν και διαφορετικά κλίματα και διαφορετικά κτίρια. Δεν είναι εύκολη δουλειά λοιπόν για μας, ωστόσο βέβαια μέσω της ανάπτυξης πρακτικών οδηγιών προς τα κράτη-μέλη και το πώς θα εφαρμοστούν στον τομέα αυτό πρακτικά μέτρα, θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό, προσπαθώντα να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται υπόψη. Είναι επίση γεγονό ότι υπάρχει ένα νέο πλαίσιο που έχει τεθεί και μια νέα οδηγία αποτελεσματικότητα ενέργεια που προβλέπει, απαιτεί από τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την διαθεσιμότητα ελέγχων υψηλού επίπεδου στους ε, ε, πολίτες και τονίζουμε ότι η υποστήριξη στον τομέα θα πρέπει να είναι υπό τον όρο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Δεν προτείνεται να υπάρξει αυτό ε, ως υποχρεωτικό μέτρο, αλλά η πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τη νέα δυνατότητα του κανονισμού για τα διαθροτικά ταμεία και το, τα δύο ταμεία επενδύσεων και να χρησιμοποιήσει τις προϋποθέσεις του να εξασφαλίσει ότι οι τομεί αυτοί και οι απαραίτητε προποθέσει υλοποιούνται από τα κράτη-μέλη και τι περιφέρειε. Δουλεύουμε λοιπόν από κοινού για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν δράσει που θα ληφθούν για να βελτιώσουν τι συνθήκε σε συγκεκριμένο τομέα. Επίση, να πω εν γέννη, διότι υπάρχει σύσταση ε, δικτών επίδοσης, ε, κάτι που θα προσέξουμε ιδιαίτερα στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Υπάρχει ένα πλαίσιο αποδόσεις που επί το οποίο υπάρχει συμφωνία. Εμείς ετοιμάζουμε τις πρακτικές οδηγίες στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας και της αποτελεσματικότητας ενέργειας να αναπτύξουμε ένα σετ δικτών επίδοσης με προσεγγίσεις καλύτερης μεγενεργειακής απόδοσης και κύκλου ζωής, φροντίζοντας ότι ο στόχος είναι να μετρήσουμε το αποτελέσμα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Να τονίσω επίσης ότι θα έπρεπε να δούμε σε ευρύτερο πλαίσιο της επενδύσης στον τομέα αυτό, διότι έχει αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, στις κοινωνικές συνθήκες, συνθήκες στα κράτη-μέλη Μερικές φορές δεν μπορούμε να απονομονώσουμε ε, αυτό το θέμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα ευρήματα της έκθεσης αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην εισηγητή. Θα είμαι σύντομος. Δεν θέλω να πω τα ίδια, θα τα πω όμως. Τα είπε και ο κύριος Ζούμπη Τι μέτρα. Για το μέλλον και λαμβάνοντας υπόψη και αυτά που είπε η Επιτροπή, περιλαμβάνει δύο τμήματα. Απόδοση, ενεργειακή απόδοση, αναμονάδα ενέργειας. Εδώ και δουλειές και ενέργεια ναι, εξοικονομούμε, ενώ το other, το, το άλλο τμήμα είναι η βελτίωση του κτηρίου. Εμείς είδαμε επενδύσεις που στην πράξη έλεγαν ενεργειακή βελτίωση, αλλά στην πραγματικότητα ήταν διακόσμηση, περιβάλλον, κήπος, λουλούδια αυτό το κομμάτι, αυτή η κατανομή θα είναι πολύ χρήσιμη. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για καλύτερη χρήση των πόρων αυτών. Ευχαριστώ. Κλείνουμε το σημείο 10 λοιπόν. Να ευχαριστήσω και τους, και τους δύο εκπροσώπους και τις Κομισιόν και του Εγκλεκτικού Συνεδρίου. Πάμε στο σημείο 11 η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας που πάει στο Μποχούνιτσε στην Σλοβακία. Σε ό,τι αφορά τον παροπλισμό των πυρηνικών εργοστασίων. Ο Γιάννης Γκάιερ είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Του δίνουμε κατευθείαν το λόγο. Γιάννης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και αυτό σύντομα μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε. Δεν υπάρχουν ε, προβλήματα στο τι θα γίνει. Η αντιπροσωπεία είχε διαφορετική βέβαια οργάνωση στην αρχή, διαφορετικό προγραμματισμό, λόγω του ότι ήταν κοντά γεωγραφικά. Είχαμε πει να πάμε μία μέρα στη Σλοβακία μονάχα και τη δεύτερη μέρα να πάμε στην Πράγα, στην Τσεχία, για να έρθουμε εκεί σε επαφή με τις αρχές και να συζητήσουμε γιατί υπάρχει ένα πάρα, ένας πάρα ψηλό ποσοστό λαθών και ξέρουμε ότι στην Τσεχία υπάρχει μια κυβερνητική κρίση που δεν έχει αρθεί ακόμη. βεβαίως ε, υπάρχουν και ε, εκλογικές εξαρτήσεις στις οποίες δεν μπορούμε να εμπλακούμε. Υπάρχει και το πρόβλημα αυτό ότι δεν υπάρχει ε, πολιτική, δεν μπορεί να λάβει κανένα την πολιτική ευθύνη μέσα σε αυτή την ανακατοσούρα, γιατί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς με κανέναν ε, συζητήσεις, γι' αυτό είπαμε να παραμείνουμε δύο μέρες στην Σλοβακία. Ε, οπότε ε, συγχωνεύσαμε λιγάκι τα, το πρόγραμμα, αλλά εγώ είμαι ικανοποιημένο με το πρόγραμμα που έχουμε. Στη δεύτερη ημέρα λοιπόν στην ε, Σλοβακία θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους αρχές που είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή των διορθωτικών ταμείων. Νομίζω χτες έγινε μια προπαρασκευαστική συνάντηση από τους ε, δύο και ήταν παρόντες ε, και από τις δύο πλευρές εκπρόσωποι Πολύ σημαντική η συνάντηση λοιπόν αυτή και σύντομα να σας πω τι έγινε. Προς το παρόν έχουμε μία μελέτη, μία συγκριτική μελέτη για, την, για το τι γίνεται με τον παροπλισμό αυτών των τριών εργοστασίων στη Βουλγαρία, στη Λιθουανία και στην Σλοβακία. Η έρευνα αυτή γίνεται από το ε, Ινστιτούτο του Φράιμπουργκ στην ε, Γερμανία όπου υπάρχει εξαιρετική τεχνογνωσία εκεί ως εξωτερικοί σύμβουλοι λειτουργούν Συνεχίζω λοιπόν. Το, το Ινστιτούτο ΕΚΟ στην Γερμανία, στο Φράιμπουργκ, μελετά το θέμα της, του παραπλησμού αυτών των αυτών των εργοστασίων. Παρακολουθούσε και την αντίστοιχη, τον αντίστοιχο παροπλισμό ε, τέτοιων εργοστασίων στο Μπράντεμπουργκ. Και το, η απάντηση ήταν ότι ναι, οι αρχές είναι σε καλό δρόμο. Παρ' όλα αυτά το πρόγραμμα δεν είναι αρκετά λεπτομερές για τον παραπλησμό, οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο όλοι οι κίνδυνοι οικονομικής ε, φύσεως ή τεχνικής φύσεως μπορούν να αναγνωριστούν, να καταγραφούν, να αξιολογηθούν και βεβαίω μπορεί να υπάρχουν και οικονομικέ συνέπειε από όλο αυτό. Το είδαμε να συμβαίνει στη Λιθουανία. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει στο Μποχούνιτσε. Δύο ώρε θα είμαστε εκεί στο εργοστάσιο, θα είμαστε με του εμπειρογνώμονε, θα συζητήσουμε, υποθέτω ότι είναι αρκετέ. Επίσης, ε, είναι αρκετά σημαντικό ο χρόνος για να ταξιδέψουμε, γιατί θα φύγουμε από τη Βιέννη και θέλουμε δύο ώρες με το λεωφορείο για να φτάσουμε. Το απόγευμα θα έρθουμε σε επαφή με μια ομάδα εκπροσώπων ε, του, της κυβέρνησης στην Πρατισλάβα, όπου ε, θα είναι ε, θα παρόντες εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Οι αρμόδιες λοιπόν κυβερνητικές αρχές που είναι υπεύθυνε για τον παρολυνικλισμό θα είναι παρόντες έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το πώς βλέπουμε εμεί την κατάσταση, πώς τη βλέπουν οι ίδιοι και αν θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνο που πρέπει να μα επισημάνουν. Και έχουμε βεβαίω πολύ συγκεκριμένα ραντεβού με το ελεγκτικό συνέδριο τη Σλοβακία. Και αυτό για μένα ήταν αρκετά σημαντικό για να έχουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για το πού υπάρχει το πρόβλημα και πώς πάει το πράγμα. Τις πληροφορίες μας τις καλύτερες τις έχουμε λάβει από το ελεγκτικό συνέδριο. Επίσης, θα δούμε τι γίνεται με τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων στην Σλοβακία. Χτες είχαμε μια συμβολή από το Γραφείο για την Περιφερειακή Πολιτική της ε, ε, Κομισιόν για τη Σλοβακία και τα ειδήσει είναι ότι η Σλοβακία ανήκει, μα δεν ανήκει στον ε, κύκλο των χωρών που είναι πολύ άσχημη η διαχείριση των περιφερειακών ε, κονδυλίων. Είναι, πολύ, είναι πάνω από το μεσόωρο, εν πάση περιπτώσει, η Σλοβακία. Βεβαίως πρέπει να δούμε πού βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα και είναι καλό να γίνει αυτό ε, σε, πίσω από κλειστέ πόρτε με την Κομισιόν, ε, με του προσώπου, για να μην μπορούν να φύγουν και και να μπορεί κανεί να λάβει τι απαντήσει που θέλει. Για να είναι λίγο τα πράγματα ξεκάθαρα. Είναι λοιπόν, ε, είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος, είμαστε όλοι για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να δεχτούμε το πρόγραμμα ως έχει, είναι αρκετά καλό. Αυτά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα είναι μικρή η αντιπροσωπεία που θα πάει εκεί και χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Γκάιερ. Παρατηρήσει υπάρχουνε. Ναι. Ο κύριος Ρούμπιχ. Δεν μπορώ να είμαι παρόν στην αποστολή, αλλά θέλω να, να θέσω ένα ερώτημα για, τον, ε, για το κόστος του ε, κύκλου ζωής ενός τέτοιου εργοστασίου. Από την πρώτη ε, μέρα που θα λειτουργήσει μέχρι τον απαροπλισμό του. Σε ό,τι αφορά την, τους παρόχους ενέργειας, τι ποσό καταβάλλεται, από τους χρήστες της ενέργειας τι ποσό καταβάλλεται, να η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης τι ποσό καταβάλει, θέλουμε να δούμε γενικώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόσο κοστίζει ο παροπλισμός, αλλά και σε εθνικό επίπεδο πόσο του κοστίζει τελικά. Καθώς επίσης και στου παρόχους ενέργειας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να θέσουμε και να είναι και διαφανή τα πράγματα. γιατί υπάρχουν και οι ε, προενταξιακές συζητήσεις και οι συνθήκες. Ε, καλό θα ήταν να τα δούμε τα θέματα αυτά. Η κυρία Μποσμπάτα. Ε, Έχουμε, εξαιρετικά καινούργια κυβέρνηση. Και υπάρχει θέμα συνταγματικό Αλλά παρόλα αυτά θα θεωρούμε ότι θα πάρει ψηφιστοσύνη στο Κοινοβούλιο. vielen Dank. Ευχαριστώ. Από την Κομισιόν να δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ. Ο Αουρέλιο Σεσίλιο, καλώς ήρθατε. Θα μπορούσατε να μας πείτε την άποψη της Κομισιόν. Is it working? Η Κομισιόν. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρούμε πάρα πολύ θετική την ε, σημασία που δίνεται σε αυτό το ε, σύστημα ελέγχου των νομοτοοικονομικών στη Σλοβακία. Θεσπίστηκε αυτό το 2004 που προσεχώρησε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά όλες τις ενέργειες κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάποιες ε, συστημικές αδυναμίες ακόμα. Μερικές από αυτές είναι ενδημικού χαρακτήρα παρά τις προσπάθειες εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Οπότε και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι έχουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και θα τονιστεί στις Σλοβακές Αρχές το πόσο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να γίνει κάποιο είδους Αναδόμιζε στο σύστημα ελέγχου και σύστημα διαχείρισης. Ιδίω τώρα που πλησιάζουμε ε, στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού του Διευθυντικών Ταμείου 2014-2020. μας κάθε βοήθεια πολύτιμη. Ενημερώσαμε το Κοινοβούλιο για το πώς έχουν τα πράγματα, ιδίως όσον αφορά το Κοινωνικό Ταμείο εδώ το είμαστε και αρμόδια, αλλά τέλος πάντων η ίδια κατάσταση σε όλα τα ταμεία. Το θέμα είναι βέβαια ότι εγώ με τις διαστάσεις του ταμείου τόσο πιο σημαντικό είναι και το πρόβλημα. Περιφερειακή ανάπτυξη, ταμείο συνοχής, ε, αντιστοίχως. Όμως, υπάρχει πρόβλημα με την ε, επιλογή και την ισότητα μεταχείριση. Προβλήματα με δημοσίε συμβάσει, προμήθειε, διαχείριση και δράσεις επαλήθευση. Αυτές είναι, αυτή είναι η βασική τομή των ε, προβλημάτων και αδυναμιών. Επίση. για τι δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες έχουμε πρόβλημα λόγω της εμπλοκής που εκείνος ότι θα έχει η δημόσια υπηρεσία των ε, ε, προμηθειών. Κατά τα άλλα θα υπαγρυπνούμε ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα έχουμε σύστημα πιο στεγανό, πιο αποτελεσματικό. Ε. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο και πάλι στο Γένσαν τον επιθυμεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ για την πρόταση που κάνετε. βεβαίω θα την ε, υποβάλουμε την ερώτησή σα. Ίσως να μην, ήταν, να μην το ε, είχαμε υπόψη μας αυτό που είπατε. Πρέπει να υπήρξε κάποια αλλαγή στην ιδιοκτησία. Ο, διευθυντής ε, τώρα, ε, μάλλον ε, ο, συγγνώμη, το, εργοστάσιο τώρα είναι κρατικό, έγινε αλλαγή της ιδιοκτησίας, οπότε θα δούμε, βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και με τα ο και με τα μέτρα. Και βεβαίως στον χρόνο που χρειάζεται πόσα ακόμα κονδύλια αναμένονται. Είναι σημαντικό αυτό Νομίζω ότι θα είναι λίγο επικίνδυνη αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα για να... γιατί αυτό το θέμα του παροπλισμού ε, θα μπορούσε να μπει στο επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, από το 2020 και μετά. Εντάξει, οι εμπειρογνώμονες λένε μπορεί κανείς να θέλει οτιδήποτε, αλλά ό,τι θέλει δεν γίνεται και πραγματικότητα. Το Μποχούνιτσο νομίζω ότι ε, έχει προχωρήσει όσο, πολύ περισσότερο από άλλα στην, στον παροπλισμό. Και οι ειδικοί λένε ότι αν είμαστε τυχεροί μέχρι το 2025 θα έχει τελειώσει. Οπότε αυτό βεβαίως θα παραμείνει στα οικονομικά μας, θα μας πιέζει για κάποια χρόνια ακόμη. υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται, κάποια που δεν γίνονται και πρέπει και εμείς να είμαστε ε, πολύ προσεκτικοί. Πρέπει όλοι να το έχουμε υπόψη. Αυτά είναι παρόδο και όπως είπα τι γίνεται με τους παλαιούς ε, ιδιοκτήτες και πού είναι το κόστος ε, και τι γίνεται με το κόστος στον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά θα τα θέσουμε. Θα δούμε τι γίνεται, τι πληρώνει το σοβατικό κράτος και οι καταναλωτές επίσης. Είναι σημαντικά τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ και την Κομισιόν. Κατάλαβα αυτό που είπε. Γι' αυτό και θα μείνουμε και άλλη μία μέρα στην Σλοβακία για να συζητήσουμε με τις αρχές για να μας πούνε τι γίνεται με τις δημόσιες προμήθειες. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι όλοι είναι αθώοι, ε, ίσως να είναι πολύ αισιόδοξη η προσέγγιση μας ως προς τις δημόσιες προμήθειες. Οι δημόσιες προμήθειες ερμηνεύονται ως ε, μια αγορά που είναι πολύ μικρή, ε, προστατεύονται οι εθνικοί ε, συμμετέχοντες, θα τα διαρευνήσουμε όλα αυτά. Θα προσέξουμε λοιπόν. Και περιμένουμε ότι όλα αυτά θα κυλήσουν καλά. Ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε μάλλον στο τέλος της ε, σημερινής συνεδρίασης. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 17 Σεπτέμβρη, στις 16 ε, και 17 Σεπτέμβρη, 3 το μεσημέρι και 9 το πρωί. Να ευχαριστήσω όλους, τη Γραμματεία, το Ελεκτικό Συνέδριο, ο πρώτος Ευχαριστή και τους Δερμηνείς και εμείς. Κλείνουμε τη συνεδρίαση σε λίγα λεπτά μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα συνεχίσουμε τους, ε, τις συνεδρίες των συντονιστών που την είχαμε διακόψει το πρωί. Σας εύχομαι σε όλους ε, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και θα χαρώ να σας δω στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. So.